Οι αρμόδιε τώρα επιτροπέ διαβίβασαν την ακόλουθη διόρθωση τροποποίηση σε ένα κείμενο το οποίο ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σύμφωνα με το άρθρο 231, παράγραφος 4 του κανονισμού μας, η τροποποίηση αυτή θα ορεθεί ότι εγκρίνεται εκτός και αν μέσα σε 24 ώρες από την ανακοίνωση μια πολιτική ομάδα ή ένας ελάχιστος προβλεπόμενος αριθμός ευρωβουλευτων ζητήσουν διεξαγωγή ψηφοφορίας. Η τροποποίηση αυτή είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας και ο τίτλος της θα κοινοποιηθεί στα πρακτικά